Ακόμα και αν εμείς ε, είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι χρειάζεται. Και πάλι εδώ μπορεί να υπάρξει μια συμμαχία μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων, γιατί ε, εγώ και να το θέσω αυτό το ζήτημα δεν έχω αρκετή επιρροή για να το προωθήσω. Η σημερινή συζήτηση είναι μια καλή αφιτηρία για να εργαστούμε από κοινού σε ό,τι αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ολοκληρώσουμε, ακολουθεί η εισηγήτρια. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Μπορέλ, για όλες τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Θα ήθελα για μια φορά ακόμη να αποτελέσω τη φωνή όσων ε, μίλησαν σήμερα και όσων εκφράστηκαν μέσω αυτής της έκθεσης σε σχέση με τα όσα προσθέθηκαν, ε, θα ήθελα να τονίσω κάποιες δυσκολίες που αναφέρθηκαν. Το θέμα του πολυμερισμού, της πολυμέρειας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό αποτελεί τον πυλώνα ε, για ε, την προώθηση των δικαιωμάτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, οι ΛΟΑΤΚΙ ε, αντιμετωπίζουν πολλέ δυσκολίε. Έχουμε και το θέμα της ε, βίας ε, κατά των παιδιών και των κοινωνικών. Επίσης, το θέμα των επιχειρήσεων που δεν αναλαμβάνουν τι ευθύνε τους, καταναγκαστική γάμη. Όλα αυτά μεταξύ πολλών άλλων είναι αυτά που θέλω να τονίσω, όπως υπόθηκαν απόψε. Κύριε Μπορέλ, ε, κατονομάσατε και τα εργαλεία, έχουμε τις αποστολές παρατηρήσεις των εκλογών, έχουμε και τη δική σας δράση. Εσείς ε, είστε είπατε εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ε, ελευθερία της θρησκείας. Όμως θα θέλαμε να αναφερθούμε και σε αυτά που μας ζητάτε εσείς καθόλου όλες διαπραγματεύσει. διαπραγματεύσεις, όσο εργαζόμαστε στην έκθεση αυτή, διάφορα πράγματα επανέρχονταν. Και είναι το εξή ένα από αυτά, ότι δεν θα πρέπει άνθρωποι που είναι ένοχοι να μείνουν ατιμόρυτοι. Θα πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον τους. Θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να επιμείνουμε επί της ε, πολυμέρειας. Θα πρέπει να επιμείνουμε έτσι ώστε το εμπόριο, ο επιχειρηματικό κόσμος να λειτουργεί με έναν τρόπο που να μας κάνει περήφανους. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στο μηχανισμό παρακολούθησης που θα έπρεπε να υπάρχει όταν ε, μιλάμε για το εμπόριο. Γιατί ε, το ένα είναι να ζητάμε κάποια πράγματα στα λόγια και είναι διαφορετικό να έχουμε και ένα μηχανισμό παρακολούθησης. Ε, έτσι, λοιπόν, ε, ελπίζω μέσα από τη θέση τη δική μας ε, εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και εσείς από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στο να συμφθεί πρόοδο στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. ενώ περνάμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Μπορέλ μπορεί να αλλάξει σελίδα. Περνάμε λοιπόν στην κοινή συζήτηση. Δηλαδή την ΚΕΠΑ και την ΚΕΠΑ. Έχουμε λοιπόν τους συζητητές, ε, τον κύριο Μακάλιστερ και τον κύριο Ντανζάν. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο και με την μπλε κάρτα και με το ηλεκτρονικό σύστημα. Και έτσι αλλάζει πλευρά ο κύριος Μπορέλ και ερχόμαστε στον ε, κύριο Μακάλιστερ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με την φετινή έκθεση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, θεωρώ ότι και πάλι έχουμε τονίσει τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πιθανές διεξόδου. Οι δύο πρώτες εβδομάδες του νέου έτους μας υπενθύμησαν ότι το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο απρόβλεπτο πιο περίπλοκο από οποιαδήποτε στιγμή από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά. Να τονίσω τρία ευρήματα της εκθεσής μου. Πρώτον, κινδυνεύει το πολυμερές σύστημα. Σε τόσο δύσκολες στιγμές όπου αμφισβητείται το πολυμερές σύστημα, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτήν την τάση και να το θέσουμε στο επίκεντρο των προσπάθειών μας για την επίλυση των συγκρούσεων. Η ΚΕΠΑ πρέπει να προωθεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις αξίες μας στη γειτονιά μας και στον κόσμο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το νέο πολιτικό κύκλο των θεσμικών οργάνων μας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πυλώνα της ΚΕΠΑ. Στην προηγούμενη θητεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στη μεσολάβηση και στην ειρηνική επίλυση διαφορών. Επιτύχαμε, παραδείγματο χάρη στην Ουκρανία και στην Βόρεια Μακεδονία. Οι προσπάθειε αυτέ. ειδικά στο πλαίσιο του διαλόγου Ζαν Μονέ, πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητά μα τα επόμενα χρόνια. Πρέπει επίση να ενισχύσουμε τον ρόλο μα στην υποπτία τη ΚΕΠΑ, αλλά βεβαίω και στα εξωτερικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να έχουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση, μεγαλύτερη συνοχή συνέπεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των εξωτερικών όργανων μας και της ΚΕΠΑ. Τρίτον, η ενίσχυση της ΚΕΠΑ για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων απειλών. Είμαι παραδείγματος χάνει πεπισμένος πως η ειδική πλειοψηφία θα καταστήσει την ΚΕΠΑ πιο αποτελεσματική και θα επιταχύνει την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ανάγκη ομοφωνίας σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δράσουμε αξιόπιστα στην διεθνή σκηνή. Όσον αφορά την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητα αυτόνομης δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συνεργασίας με περιφερειακούς οργανισμούς. Η ανακοίνωση της Προέδρου της Κομισιόν για μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση τα επόμενα πέντε χρόνια είναι ευπρόσδεκτη. Τέλος, συνάδελφοι. Κανένα κράτο μέλο δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στι παγκόσμιε προκλήσει από μόνο του. Πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε τι ευρωπαϊκέ αξίε μα παραμένοντας προσιλωμένοι σε μια διεθνή τάξη που θα βασίζεται σε κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλο παίκτη όταν μιλάμε για την διπλωματία, το εμπόριο, την αναπτυξιακή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και βήμα-βήμα και στον τομέα τη ασφάλεια και άμυνας η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει στρατηγικά χρησιμοποιώντα τι πολλέ πολιτικέ που έχει στη διάθεσή τη για να ανταποκριθεί στις προκλήσει στη γειτονιά μα και παραπέρα. Είναι και καινή ώρα για να πάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας και να εμφανιστούμε ως μια κυρίαρχη οικονομική και πολιτική δύναμη στις διεθνείς σχέσεις. Και θέλω να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο ύπατος εκπρόσωπος της πρώτης εβδομάδας. Νομίζω ότι έχει τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Τέλος, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας για τις ε, συνεισφορές τους, ε, ιδίως τους σκιώδεις για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντανζάν, εισηγητής της δεύτερης έκθεσης. Επιτρέψτε μου Καταρχήν να ευχαριστήσω ειλικρινά το σύνολο των σκιωδών εισηγητών, ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας και ανεξαρτήτων των διαφορών μας. Όλοι προσπάθησαν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ετήσια έκθεση. Είχαμε αρκετά απαθιασμένο διάλογο, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, για αυτό το θέμα. Κατά την άποψή μου μπορούμε να κάνουμε μια ρεαλιστική διαπίστωση ε, για τα θέματα της ε, άμυνας και για τη δυνατότητα βελτίωσης. Τουλάχιστον σε αυτό το πνεύμα εκπώνησε αυτή την έκθεση που τροποποιήθηκε αρκετά. Ο ρεαλισμός στη διαπίστευση είχε να κάνει με την επιδίνωση του κλίματος ασφάλειας. Έχουμε σειράξεις στη Λιβύη, στη Συρία, στην Ουκρανία, ε, τζιχαντιστικές επιθέσεις, ε, έχουμε ε, και στο Σαχέλ, ανατεραχή, ακόμη και στην Ευρώπη. Έχουμε ταυτόχρονες κρίσεις, αλληλένδετες και βλέπουμε αξιοθρύνητες εικόνες μιας Ευρώπης σχετικά αδύναμης. Η ιδιαίτερη αστάθεια της κατάστασης έχει ανατρέψει τις βεβαιότητές μας καθώς ε, ε, και είναι και ε, μεταβλητές και οι συμμαχίες μας. Έχουμε το παράδειγμα στη Μέση Ανατολή. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ότι πέρασαν τα άσχημα, ίσως, ίσως και όχι και ε, τι να πω, μάλλον όχι. Μου φαίνεται σήμερα ότι είναι ανεύθυνο, ενώ είμαστε Ευρωπαίοι, να σκεφτόμαστε ότι η ασφαλειά μας θα συνεχίζεται ε, να διασφαλίζεται αιωνίως από άλλους, χωρίς να κάνουμε σημαντική προσπάθεια να αναλάβουμε τις ευθύνε μας. Έτσι. Λοιπόν, ο λυσμός της διαπίστευσης είναι ότι υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή εποτυχία και θα πρέπει ε, να ε, έχουμε ρεαλιστικές συστάσεις για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να δράσουν επιτέλους και όχι απλώς ε, να καταδικάζουν. Τα κράτη-μέλη είναι και θα μείνουν ουσιαστικοί πρωταγωνιστές στον τομέα της άμυνας. Όμως είναι ρεαλισμός να γνωρίσουμε ότι κανένα εξ αυτών ούτε και το πιο φιλόδοξο και σας το λέει ένας Γάλλος δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ε, και ε, βλέπετε τι έγινε στο Σαχέλ, ε, είπατε εκπρόσωπε. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή συνεργασία και θα πρέπει να έχουμε υποστήριξη στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να έχουμε ε, ε, μόνιμες δομές, όμως αυτές δεν θα έχουν ακόμη και μεσοπρόθεσμα σημαντική διαφορά. Έτσι λοιπόν πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε ικανοποιημένοι που είμαστε απλώς ε, θεατές ε, και μερικές φορές ακόμη και ζητιάνοι ε, της παγκόσμιας ασφάλειας απέναντι σε παγκόσμιες δυνάμεις. Θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές και να έχουμε τα μέσα. Ξέρω τι γίνεται με τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία, αλλά θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Καταρχήν πρόκειται για μια φιλοδοξία προς μισή και όχι μια απόλυτη πραγματικότητα σήμερα. Ε, δεύτερον, τον ε, το να είναι αυτόνομο κανεί δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει τι συμμαχίε και τι συμπράξει, αλλά θα πρέπει να αξιολογεί τι καταστάσει κρίση από μόνο του και να μπορεί, αν χρειαστεί, να απαντήσει μόνο του, δίνοντα μία απάντηση που θα σέβεται τι δικέ μα προτεραιότητε. Το να διαπιστώσουμε οι προτεραιότητε τη ασφάλεια για εμά, ο Ευρωπαίου, δεν είναι ακριβώ ίδιες με τις προτεραιότητες ε, ε, των συμμάχων μας εκτός της Ευρώπης ε, δεν είναι μια αντιπραστική αρρώστια. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Συζητάμε πάρα πολύ για τα κλιματικά θέματα, για τα κοινωνικά θέματα στο κύκλο. Νομίζω όμως ότι είναι επίγον να εργαστούμε και να αξιολογήσουμε το θέμα της στρατηγικής μας θέσης. Ακολουθεί ο ύπατος εκπρόσωπος. Κύριε Μπορέλ Φοντέλες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μακάλιστερ και τον κύριο Νταντζόν για όλα όσα έχουν κάνει, προετοιμάζοντας αυτές τις ε, εκθέσεις για την ε, ΚΕΠΑ και την ε, ΚΑΠΑ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να μιλήσουμε για την ε, συνέχεια που θα δώσουμε στον κεντρικό χαρακτήρα αυτών των αξιών. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μία δύναμη που βασίζεται σε αξίες. Η πολυμέρεια και μία διεθνής ε, τάξη βάση κανόνων αποτελεί τη βάση της εξωτερικής μας πολιτικής με τα χαράς βλέπω να γνωρίζετε ότι πρέπει να είμαστε ε, πιο δυναμικοί. Και έχουμε σήμερα την απόδειξη ακριβώς αυτού σε σχέση με τη Λιβύη και με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί λοιπόν στην προστασία των ζωτικών μας συμφερόντων. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου ε, η πολιτική καθορίζεται με βάση την εξουσία και χρειαζόμαστε λοιπόν μια εξωτερική πολιτική που ε, συνδυάζει την εξουσία και την ισχύ μάλλον των ε, κρατών μελών μας με την ε, συνεργασία μεταξύ μας. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την διασύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Αυτό έχει υποθέσει πολλές φορές, καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε. Καλύτερα ακόμα θα ήταν να το υλοποιήσουμε χαιρετίζω την έμφαση που δίνεται στη σημασία της διασφάλισης επαρκών δημοσιονομικών πόρων για την εξωτερική δράση υπό το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα εξετάσουμε σύντομα και θα δούμε αν αυτό είναι δυνατόν ή όχι. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να διατηρήσουμε τα χαρτοφυλάκια για την υποσαχάρια Αφρική, την πολιτική γειτονία στο νέο μηχανισμό. Χθες ε, συνάντησα τον μεγάλο Πρόεδρο και το, τους Προέδρους των πέντε χωρών της Ποσαχάριας Αφρικής. Και το ζήτημα των πόρων που απαιτούνται για να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουμε και εμείς, είναι λοιπόν ένα θέμα που ε, ετέθη επιτάπητο και δεν ξέρω κατά πόσο η απάντηση που θα του δώσουμε τις επόμενες ημέρε είναι επαρκής. Η πολιτική. Τώρα, πολύ σωστά είπατε ότι ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε χρειαζόμαστε εταίρου. Θέλουμε την πολυμέρεια, αλλά για την πολυμέρεια απαιτούνται και άλλοι. Δεν φτάνουμε μόνο εμείς. Για τις διμερείς σχέσεις χρειαζόμαστε δύο, για τις πολυμερείς χρειαζόμαστε πολλούς. Θέλουμε ε, εταίρους όπως ε, ε, την Αφρικανική Ένωση, τον ΟΗΕ και άλλους. Αν δείτε για παράδειγμα την κλιματική αλλαγή, στην τελευταία συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συζητήσαμε πώς θα αναπτύξουμε μια ισχυρή πολιτική διπλωματία προκειμένου οι περιβαλλοντικές μας φιλοδοξίες να μπορούν να προαχθούν σε συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε μαζί με άλλους, να τους ε, πείσουμε για τις κλιματικές μας ε, δράσεις, προκειμένου αυτές πραγματικά να πετύχουν το στόχο τους. Αξιοπιστία. Είναι σαφές ότι ε, πλήττεται η αξιοπιστία μας ως γεωπολιτικής δύναμης εάν δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας ό,τι αφορά την σταθερότητα και την ειρήνη στην άμεση γειτονιά μας. Ε, να τουλάχιστον αν δεν λύσουμε τα ζητήματα, τουλάχιστον να βοηθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα των Δυτικών Βαλκανίων και τη Λιβύη. Αλλιώ θα είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε κάποιον ότι είμαστε ισχυρή πολιτική δύναμη. Αυτό είναι σαφέ και θα πρέπει να αυξήσουμε την ε, στήριξή μα ε, προ την εθνική κυριαρχία ε, Μίλησα για το κοσμοπέδιο. Ακόμα δεν ε, μπορούμε να πάμε γιατί δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα, θα πρέπει να πάμε στο κοσμοπέδιο και τη Σερβία προκειμένου να επαναλάβουμε την ε, προσήλωσή μας προς, το, προς την ευρωπαϊκή προσέγγιση και όραμα για όλη την ευρύτερη αυτή περιοχή. Υπάρχουν δυσκολίες με κάποιους από τους γείτονές μας. Οι πρόσφατες δράσεις ε, της Τουρκίας ε, δημιουργούν ε, προβλήματα στις σχέσεις μας. Η Κεντρική Μεσόγειος περνάει από τρομερές αλλαγές από γεωπολιτικής άποψης. Κάποιοι φορείς όπως η Ρωσία και η Τουρκία πριν από έξι μήνες δεν είχαν καμία παρουσία εκεί. Τώρα βλέπουμε ότι βγαίνουν μπροστά. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγάλη προσοχή προς τα δεξιά μας, αλλά και προς ε, τον Νότο, ε, Λιβύη, Ιράν, Ιράκ, που βρίσκονται στο προσκήνιο σήμερα. Βρισκόμαστε στην ε, πρώτη γραμμή των προσπαθειών προς την αποκλιμάκωση, όμως τελικά πρέπει να δούμε ε, ποιο κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και διαπραγματεύεται την εκεχηρία. Δεν είμαστε εμεί, αλλά η Ρωσία και η Τουρκία. Αφρική. Α μιλήσουμε για την Αφρική. Ε, μία πολλά υποσχόμενη ε, ήπειρο που αντιμετωπίζει και σημαντικέ προκλήσει όμω. Υπάρχει εντολή από το Συμβούλιο προ την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να παρουσιάσει μέχρι τον Ιούνιο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τον Ιούνιο για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πλάνο ε, για την Αφρική. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να καταρτήσουμε ένα σχέδιο για την Αφρική χωρίς τους Αφρικανούς. Ξεκινώντας από το Σαχέλ, ο πρόεδρος Μακρόν χθες είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους προέδρους των πέντε χωρών της του Σαχέλ και τους ζήτησε να πούν τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς στην Αντίσα Μπέμπα το Φεβρουάριο. Λατινική Αμερική. Φλέγεται από την Χιλή μέχρι το Μεξικό. Έχουμε πολλές και σημαντικές δυσκολίες εκεί και θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία μας για να προωθήσουμε τα συμφέροντα μας στην Ασία, που είναι ε, ευημερούσα και σταθερή, ίσως η πλέον σταθερή και ευημερούσα περιοχή του κόσμου σήμερα. Θα ε, μεταβώ στον Δελχή αύριο για να συμμετάσχω στον διάλογο εκεί και να, και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Το ίδιο θα πράξω σύντομα και με την Κίνα, ε, προετοιμάζοντα την Σύνοδο Κορυφή. Για την ε, ΚΕΠΑ τώρα και την σχετική έκθεση που αντιμετωπίζει την ε, σημαντική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Εδώ είναι σαφές το μήνυμα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλη επιλογή από το να ενισχύσει τι ικανότητε τη για να προστατευθεί και να αποτελέσει έναν πιο αξιόπιστο πάροχο ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 17 επιχειρήσεις ε, πέραν των συνόρων μας. Και χαιρετίζω τον ενθουσιασμό και την αφοσίωση χιλιάδων ανδρών και γυναικών που υπηρετούν ε, και περασπίζονται την ευρωπαϊκή σημαία, ορισμένες φορές υπό επικίνδυνες συνθήκες. Στην έκθεσή σας, σωστά επισημαίνεται ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, συστηματικά, δομικά ζητήματα που μας πλήττουν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις ε, της ΚΕΠΑ θα γίνουν πιο εύρωστες από πλευράς ανθρωπίνων πόρων και από πλευράς εντολής. Χαιρετίζω την πολιτική στήριξη για τη δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής Ειρηνευτικής Δύναμης εκτός προπολογισμού. Αυτό θα επιτρέψει στους εταίρους μας ε, να ε, διαφυλάξουν την ασφάλειά τους δημιουργώντας τις δικές τους ικανότητες. Αυτό ισχύει στην υποσαχάρια Αφρική συγκεκριμένα. Πρέπει να αναπτύξουμε στρατηγική αυτονομία ένας όρος ε, που ερμηνεύεται διαφορετικά ανάλογα με το που στέκεται ο καθένας. Είναι ε, λεπτό το ζήτημα. Σε αυτό το πλαίσιο όμως αυτός ο όρος σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητά μας ε, να συνεργαζόμαστε με τέρους όπου αυτό είναι απαραίτητο ή και μόνοι μας αν αυτό είναι απαραίτητο. Στην έκθεσή σας αναφέρεται ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέτει κατά μέρος τις εταιρικές της σχέσεις. Αντιθέτως, αυτό θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν ισχυρότερο ε, παγκόσμιο φορέα και θα ωφελήσει και τον ΝΑΤΟ, γιατί μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα πιο ισχυρό ΝΑΤΟ ε, είναι, ε, συμβαδίζουν. Τώρα, το μόνιμο Ταμείο Συνεργασίας και στρατικής Συνεργασίας ε, εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε το ποσό που θα δοθεί σε αυτό το ταμείο, καθώς και στον μηχανισμό ασφάλειας που θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο της μελλοντικής, των μελλοντικών έργων ε, ΚΕΠΑ. Πολλά μπορούμε να πούμε εδώ για τα όσα προσπαθούμε να κάνουμε. Τα καλύπτει η έκθεσή σας ε, εξαιρετικά. Συμφωνώ με όλα όσα επισημαίνεται εκεί. Θέλω μόνο να τονίσω την σημασία των νέων συνόρων τεχνητής νοημοσύνης που θα έχουν γεωπολιτικές προεκτάσεις, ενδυναμώνοντας ε, ανταγωνιστικά μεταξύ τους ε, ε, κράτη και εχθρικούς μη κρατικούς παράγοντες. Πρέπει να παραμείνουμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο για τους κανόνες ε, καθώς και από τεχνολογικής άποψης ε, για να αναπτύξουμε τα δικά μας ε, μέσα ασφαλείας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν γνωρίζουν τη σημασία αυτού του θέματος. Ποιες θα είναι οι συνέπειες της ανάπτυξης τεχνολογιών, τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την ασφάλειά μας στο μέλλον. Και όταν λέω μέλλον, δεν εννοώ πολύ μακριά, στην επόμενη πενταετία οι εξελίξεις θα είναι καθοριστικές. Και στη θάλασσα, άλλος ένας ε, στρατηγικός ε, τομέας όπου πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, κοινή συνεργασία, συνεργασία και αξιοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών μηχανισμών. Και εδώ επισημαίνω, όπως κάνετε και στην έκθεσή σας, ότι το δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί αντίστοιχη διαρθρωτική χρηματοδότηση, ιδίω από τον Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, για να διατηρηθεί η συμβολή του στις ενέργειές μας. Είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε δράσεις σε όλο τον κόσμο εάν δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τον κόσμο. Την Ιφίλιο. Έχουμε ένα δορυφορικό κέντρο το οποίο δεν γίνεται να στερείται πόρων για να επιτελέσει το έργο του. Κλείνοντας, είναι μεγάλο το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, τεράστια η πρόκληση. Πρέπει να διατηρήσουμε τη δυναμική μας ε, για την ενίσχυση της ε, κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στην άμεση γειτονιά μας και στο άμεσο μέλλον που όπου θα πρέπει εμείς να δώσουμε δείγματα γραφής για την ικανότητά μας και για την δυνατότητα των κρατών μελών να διαμετρήσουν αυτό το ρόλο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λιβύη, για παράδειγμα. Φανταστείτε μόνο να υπάρξει εκεχηρία. Και στο Βερολίνο υπάρχει συμφωνία για την έβρεση πολιτικής ε, λύσης. Ας φανταστούμε λοιπόν ένα τέτοιο σονάριο. Μια κεχηρία δεν μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες χωρίς μια ισχυρή διαδικασία παρακολούθησης. Θα είμαστε εμείς έτοιμοι για αυτό το σενάριο, για αυτό το ενδεχόμενο. Θα πρέπει να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα στο προσεχεσμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κερδίζουν, ε, αρχίζουν τώρα οι κοινοβουλευτικέ ομάδε με τον κύριο Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από το εκτελεστικό πρώτα απ' όλα να κάνει τα του οίκου μας πριν προχωρήσει στα εξωτερικά. Στη Λιβύη, παραδείγματο χάρη, θεωρώ ότι έχουμε διαφορετικά συμφέροντα. Φροντίστε λοιπόν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να είναι συντονισμένες ε, και τουλάχιστον να διαλέξουν ε, εάν είναι στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης ε, κυβέρνησης ε, και να φροντίσουν να ασχοληθούν όσο τουλάχιστον ασχολείται και η Γαλλία με το ζήτημα και φροντίστε να μην κοπούν τα κονδύλια για το αμυντικό ταμείο και την στρατιωτική κινητικότητα. Και για να τελειώσουμε κάτι το θετικό, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα νησί στην Ανατολική Ασία όπου υπάρχει μια κινέζικη κοινωνία που κάνει δημοκρατικές εκλογές. Σας συγχαρούμε λοιπόν τον λαό της Ταϊβάν για τις εκλογές που διεξήχθησαν και αυτό ευχόμαστε για ολόκληρη την Ανατολική Ασία. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες. Ο κύριος Λόπες, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά αυτή την ολομέλεια εγκρίναμε δύο σημαντικές εκθέσεις για την εξωτερική πολιτική, την έκθεση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και την έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο ε, Μακάλιστερ για τη συνεργασία. Οι δύο αυτές εκθέσεις ε, ε, ουσιαστικά διαπιστώνουν ότι ο κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικός από τις τελευταίες δεκαετίες. Ο ανταγωνισμός μεταξύ με των μεγάλων δυνάμεων απειλεί τον τρόπο που κατανοούμε τον κόσμο, ένα κόσμο που βασίζεται σε πολυμερείς δομές και κανόνες πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να συνεργαστούμε παρά να αντιγωνιζόμαστε ε, και ότι πρέπει να δρούμε μέσω του διαλόγου. Μπροστά σε αυτή τη διαπίστωση η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει να ακολουθήσει, ε, μάλλον να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της και ε, γι' αυτό πρέπει να στοιχηματίσουμε στη δική μας αυτονομία και στη δική μας κυριαρχία ως Ήπριος για να έχουμε τις ικανότητες να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και να προωθήσουμε τα συμφέροντα και τις αξίες μας. Από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη Ευρώπη ε, είναι χορτοφαγικό όν σε ένα κόσμο σαρκοφάγων. Ε, και τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους κατάλληλους πόρους, να έχουμε νέε ικανότητες στην άμυνα, να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας, ιδίω με τη Λατινική Αμερική και την Αφρική και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας ε, και μεταξύ των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό είπε το εκπρόσωπος έχει κεφαλαιόδη ρόλο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ για το Renew Europe, ο κύριος Παέτ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, για να ακουστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα παγκόσμια ζητήματα και για να την ε, ε λάβουν σοβαρά, θα πρέπει να έχει μια νέα φωνή. Εδώ μιλάμε για τομεί εξωτερική πολιτική, αναπτυξιακή συνεργασία και διεθνού εμπορίου, καθώ και την πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Πολλά έχουν ε, γίνει στο ε, θέμα τη πολιτική ασφάλεια και άμυνα, αν συγκρίνουμε τα προηγούμενα έτη, αλλά και άλλα πρέπει να γίνουν. Και αυτή η ιδέα τη κοινή άμυνα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλα τα κράτη-μέλη. Καθώς ο στόχος είναι η στρατηγική αυτονομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της ευρωπαϊκής και της ασφάλειας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με το ΝΑΤΟ και άλλους εταίρους που έχουν τις ίδιες ιδέες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποσκαφθεί ο ρόλος ε, του ΝΑΤΟ. Το αντίθετα, μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρότερο εταίρο ε, για το ΝΑΤΟ, θα συνεισφέρει με μεγαλύτερε αμυντικέ ικανότητε, θα επενδύσει στι επενδυτικέ τεχνολογίε ή με άλλα μέσα. Λαμβάνοντα υπόψη το μέγεθο και τι ικανότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι θεμελιώδε ότι θα πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό τη. Για το λόγο αυτό, η πολύ καλή συνεργασία τον ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και άλλους είναι πολύ σημαντική. Όμως για να μπορούμε να υπερασπίσουμε τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του πολυμερού συστήματος που αποτελεί ε, τη βάση ε, της ασφάλειας και της άμυνας ευρωπαϊκής ικανότητες. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αμυντική της πολιτική θα πρέπει να έχει τα πάντα ε, στρατηγικές ικανότητες, προσωπικό και τεχνολογικές ικανότητες ε, μέχρι αποτελεσματική αμυντική βιομηχανία. Απαιτούνται οι επαρκείς ε, πόροι καθώς και να υπερβληθούν οι πολιτικές διαφωνίες. Διαφορετικά δεν θα έχουμε λόγο δίπλα σε άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως είπα η Κίνα και άλλοι. Έχουμε κάποιες άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να δώσουμε ήδη προσοχή και να τις αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε τον κύριο Κόφερ για τους πράσινους. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Ζαν Κλωτιούκερ μίλησε για δυνατότητα άσκησης παγκόσμιας πολιτικής. Αυτό είναι το επίκεντρο της ΚΕΠΑ. Και συμφωνώ κύριε Μπορέλ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εψυχάζουμε στο status quo. Πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε νέες προκλήσεις. Βεβαίως, πρέπει να έχουμε ξεκαθαρή κατεύθυνση. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας χωρίς να πέσουμε στην παγίδα της μεγάλης δύναμης. Να μην γίνουμε τρίτη υπερδύναμη, αλλά να μην υποταχθούμε και στις υφιστάμενες Γι' αυτό πρέπει να αποτελέσουμε πυλώνα μιας πολυμερούς τάξης και να συνεισφέρουμε για να ισχύσει διεθνώς το δίκτυο και να μην αποτελεί μια ανάμνηση παλιά. Η έκθεση του κυρίου Μακάλιστερ είναι μια καλή έκθεση και σας ευχαριστώ γι' αυτό και ελπίζω να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και με τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων και να συνεννοηθούμε. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Μπον Φρίσκο για την ομάδα ID. Μικρόφωνο παρακαλούμε για την ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τους συζητητές Μακαλιστέρ και Ντανσάν για την εξαιρετική δουλειά τους και για τις εκθέσεις τους. Εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε πόσα λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική ε, έχουν υλοποιηθεί χωρίς ε, να έχει ε, συνεισφέρει στην επίλυσή τους ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα βλέπουμε ότι η Λιβύη κλειστά στα χέρια της Ρωσία, της Τουρκία ε, και τη Κίνα Ενώ με την πρώτη δυσκολία εγκαταλείπουμε τη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Όμω η απλή ερώτηση, κύριε Μπορελή, τα πολιτικά μέσα και οι πόροι για την αμυντική βιομηχανία θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο ασφάλειας για τους Ευρωπαίους πολίτες που εκλέγουν αυτό το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί για το ECR ο κύριος Φανόρντεν. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ανήκα στους λίγους συντηρητικούς που είχαμε εκλεγεί το 1999 που προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις πραγματικές ανησυχίες και φιλοδοξίες των πολιτών μας. Για μια κοινή αγορά αντί για τις ομοσπονδιακές ε, ιδεολειψίες μιας μικρής ελίτ και για να προστατεύσουμε την εθνική μας ε, κυριαρχία. Στον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας είναι οι ένοπλες δυνάμεις, οπότε βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τις ελέγξει. Αναγνωρίζω επίσης πως κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες πρέπει να είναι η δέσμευση των ΙΠΑ για την ασφάλειά μας μέσω του ΝΑΤΟ. Οι ανησυχίες μου για αυτά τα ζητήματα ήταν ο λόγος για τον οποίο ήμουν κατά της ε, ΚΕΠΑ, του Ευρωστρατού θα έλεγαν κάποιοι, όσο καιρό βρίσκομαι σε αυτό το κοινοβούλιο. Οι εκθέσεις εδώ πέρα ζητούν ειδική πλειοψηφία για ζητήματα που θα έπρεπε να είναι εθνικά προνόμια και η στήριξη του κυρίου Ντανζάν μιλάει για στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή μακριά από τις ΗΠΑ. Χωρίς να σκέφτεται τι σημαίνει αυτό, λέει δύο λόγια για το ΝΑΤΟ, αφιερώνει μία παράγραφο στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, αναζητά μία Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, τον αποχωρισμό από τους διατλαντικούς συμμάχους μας. Δεν έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν. Όλοι πρέπει να ενισχύσουμε τις εθνικές στρατιωτικές ικανότητες μας, να είμαστε καλύτεροι σύμμαχοι και να εξηγήσουμε την ανάγκη για αξιόπιστη άμυνα στους πολίτες μας, αλλά οι δημοκρατίες πρέπει να είναι αλληλέγγυες στη μεγάλη συμμαχία του ΝΑΤΟ και να μην δημιουργήσουν εναλλακτικέ δομές που οδηγούν σε διχασμό. Υπάρχει μια μπλε κάρτα την δέχεστε. Παρακαλώ. Κύριε Βανόρντεν, δεν ήσασταν πάντα με την πλειοψηφία σε αυτά τα ζητήματα και ε, διαφωνούμε σε αρκετά. Συμφωνούμε ίσως ε, στην άποψή μας για το ΝΑΤΟ και την ανάγκη να ενισχύσουμε την διατλαντική μας συνεργασία. Θα μου επιτρέπετε να συνεχίσω να ελπίζω καθώς πρόκειται για την τελευταία σας ολομέλεια ότι θα νοσταλγείτε λίγο ε, τα χρόνια που περάσαμε μαζί και τη δουλειά που κάναμε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δέχτηκα την κάρτα σας ε, με μεγάλη ευχαρίστηση Ε, Βεβαίω σε μια προηγούμενη συζήτηση δύο συμπατριώτες μου δεν δέχτηκαν ερώτηση δική μου. Κοιτάξτε, θα φύγω από αυτό το κοινοβούλιο με κάποια θλίψη. Οφείλω να πω, πέρασα 30 χρόνια ως στρατιωτικός, 20 ε, χρόνια τη ζωή μου εδώ ως πολιτικός. Επιτύχαμε κάποια καλά πράγματα μαζί. Αλλά υπάρχει τώρα αυτή η τάση, η οποία επιταχύνεται με την Βρετανική αποχώρηση που νομίζω οδηγεί τα πράγματα σε λάθος κατεύθυνση και με ανησυχεί. Συνεχίζουμε λοιπόν με την κυρία Βίλα Νουέβα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Πρόσφατα κλιμακώση των εντάσεων που είδαμε στο Ιράν μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί έθεσε τον κόσμο σε μεγάλη ένταση. Πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες ε, αν τι είναι πολιτική Τραμπ. Ε, η ασφάλεια δεν λύνεται με στρατιωτικές επιχειρήσεις. θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις, πρόσβαση στην απασχόληση επίσης ασφάλεια είναι να μην έχουμε επεμβάσεις στρατιωτικές σε άλλε χώρες, ε, ούτε να συμμετέχουμε σε βομβαρδισμούς από ντρόν ε, ή σε επεμβάσεις του Λευκού Οίκου. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το διεθνέ δίκαιο. Πρέπει να ενισχύσουμε το πολυμερές σύστημα, όμως ε, γι' αυτό Πρέπει να έχουμε ε, το δικό μας ε, ρόλο. Βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή για την ε, ίδια την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίων. Να δώσουμε προτεραιότητα στο διάλογο, στη διπλωματία, το δημοκρατικό έλεγχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, να στοιχηματίσουμε στην ασφάλεια και στην δίκαιη ανάπτυξη άλλων χωρών, στην προστασία του πλανήτη, στο φεμινισμό και στη δημοκρατία. τότε θα υποστηρίζουμε και θα ενισχύουμε την την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδάκης έχει το λόγο για τους μη Καθαρά πράγματα. Οι δύο εκθέσεις συνιστούν προετοιμασία νέων πολέμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα της πολυμερούς αυτόνομης δράσης και της νέας γεωπολιτικής επιτροπής από κοινού ή χωρίς το νατο μεθοδεύεται η υποστήριξη των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ομίλων στον ανταγωνισμό τους με τους αντίστοιχους ομίλους αμερικάνικους κινέζικους και ρώσικους. εξαγγέλλονται περισσότερες υπερελιστικές επεμβάσεις σε τρίτες χώρες αυξημένοι εξοπλισμοί και πέραν αυτών του νατο ενώ πολλαπλασιάζονται οι ευρωνοσιακοί στρατιωτικοί μηχανισμοί κάτω από την ομπρέλα της ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης όπως η ΠΕΣΚΟ, η στρατιωτική αξιολόγηση τύπου card το ταμείο άμυνας ο μηχανισμός γειτονίας ο προκλητικά ψευδεπίγραφος μηχανισμός για την ειρήνη ως και το ευρωπαϊκό συμβούλιο ασφαλείας προωθείται. όλα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με υπεράσπιση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως ισχυρίζονται φυσικάζοντας οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. γι' αυτό άλλωστε και για το αυθαίρετο τουρκολιβικό σύμφωνο η ευρωπαϊκή ένωση δηλώνει απλώς ανήσυχη ενάντια λοιπόν στα σχέδια της συμπεριλαστική λυκοσυμμαχία της ευρωπαϊκής ένωσης οι λαοί να απαλέψουν για καμία αλλαγή συνόρων και συνθήκων που τα καθορίζουν με ξύλωμα όλων των ξένων βάσεων και μηχανισμών. Η έκθεση Κάλιστερ και η έκθεση Ντανζάν, είναι εξαιρετική οδηγή για να πάμε παραπέρα, για να δημιουργήσουμε το απαραίτητο όραμα και να δώσουμε απαντήσεις που δεν βρίσκουμε σήμερα. Θα αναφερθώ κυρίως στην έκθεση Ντανζάν, γιατί αυτό παρουσιάζει ε, ένα όραμα, έχοντας κατά νου ότι η άμυνα είναι ένας ε, εξειδικευμένος τομέας και άπτεται της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Στον τομέα της άμυνας, τα κράτη-μέλη έχουν ισχυρή εντολή και δεν ε, έχουν κοινή συνεννόηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Άμυνα έχουν ε, διάφορες ε, στρατηγικές. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει κυρία αντίληψη απέναντι στις απειλές. Ε, υπάρχει μεγάλη γκάμα απόψεων σε σχέση με τη χρήση των στρατιωτικών δυνάμεων. Ούτε υπάρχει κοινό όραμα, κοινή οπτική σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού στρατού. Το Διεθνές Ινστιτούτο για τις Στρατηγικές Μελέτες εκτιμά ότι θα χρειάζονταν περίπου 350 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς μικρόφωνο μιλτής σε ένα σενάριο ε, που θα έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό της η Ευρώπη. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο. Ξεπεράσει το χρόνο, με συγχωρείτε και ο χρόνος πιέζει. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο Άρα Κόβατς. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ε, έχουμε ένα πολύ καλό κείμενο, χάρη στον κύριο Ντανζόν, και θεωρώ ότι χάρη στι κοινέ προσπάθειε των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου, καταφέραμε να κρατήσουμε ένα εξαιρετικό έγγραφο και με τους σκιώδεις καταφέραμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Ε, συμπεριλάβαμε όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα και πολύ σημαντικά για τους Ευρωπαίους Δημοκράτες ε, και ενισχύουμε και τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Επίσης, στην έκθεση τονίζεται η σημασία και αναγκαιότητα της ε, βαθύτερης ολοκλήρωσης Όλα αυτά είναι σημαντικά στο πλαίσιο των ε, Ευρωπαϊκών ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί θεωρούμε ότι μόνο μια κοινή αντιμετώπιση μπορούμε να επιλύσουμε τα ζητήματα. Μόνο μία ενωμένη ισχυρή Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο λαϊκισμό, ε, της επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, της εκστρατείες παραπληροφόρησης. Με την έκθεση αυτή κάνουμε ένα βήμα προς την επίτευξη των στόχων και ονείρων μας. Γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω να την υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάουτμανς. Το 1999 η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε ότι είχε λύσει το ζήτημα, το ερώτημα του Henry Kissinger. Ποιον να καλέσω όταν θέλω να μιλήσω με την Ευρώπη. Δημιουργήθηκε μια νέα θέση λοιπόν του ύποτου εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων. Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι το ερώτημα του Κίσιντζερ δεν έχει επιληθεί. Βλέπουμε σήμερα με την κατάσταση στο Ιράν, στο Ιράκ, μετά τον θάνατο του στρατηγού Σολαϊμανή, ότι όλοι καλούν τους πάντες. Κύριε Μπαρέλ, εσείς ε, μιλάτε με τον ε, Ζάρεφ. Ο Μισελ παίρνει τον κουτέρε, άλλοι παίρνουν τον Ροάνι, άλλοι τον Έρντογαν. Πρέπει τα πράγματα κάπως να ξεκαθαρίσουν και να γίνουν πιο αποτελεσματικά, όχι μόνο για τους κίσιντζερ αυτού του κόσμου, αλλά για να υπερασπιστούμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Κύριε Μπορέλ, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες καταλαβαίνουν ότι εσείς είστε σαν ένας ε, Ευρωπαίος Υπουργό Εξωτερικών. Μόνο έτσι θα το κατανοήσουν όλοι. Πρέπει να έχετε ε, τα απαραίτητα εργαλεία, να καταργηθεί ε, ο κανόνας της ε, ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Ε, για να μπορείτε εσεί ε, ακόμα και σήμερα να ταξιδέψετε στην ε, Τεχεράνη ή στην Νέα Υόρκη. Να έχουμε μια πραγματική αμυντική ένωση και αν με ρωτάτε με έναν πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Αν μπορούμε κάτι να μάθουμε από τους Ρώσους και τους Αμερικάνους είναι το εξή. Μια ισχυρή εξωτερική πολιτική μαζί με έναν ισχυρό στρατό είναι το κλειδί. Πρέπει λοιπόν να παλέψουμε για μια ισχυρότερη Ευρώπη. Και κύριε Μπορέλ, εμείς θα αγωνιστούμε μαζί σας σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την κυρία Νόημαν για ένα λεπτό. Πατήστε το μικρόφωνο. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπουμε πάλι τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ε, τα περισσότερα όπλα όμως δεν κάνουν την περιοχή ασφαλέστερη. Χρειάζεται αφοπλισμός και πρόληψη. Αλλά από αυτά δεν βλέπουμε τίποτα στην έκθεση του κυρίου Ντανσάν. Δεν υπάρχει κάποια ανάλυση των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα λεφτά ζητάτε παρά το ότι εξάγουμε όπλα τα οποία ρίχνουν ε, λάδι στη φωτιά. Ανταυτού η έκθεση ζητάει να φτάσουν οι εξοπλισμοί στο 2% του ΑΕΠ. Πολλές φορές μάλιστα το επαναλαμβάνει. Εμείς όμως θέλουμε μια πολιτική ασφάλεια που θα βασίζεται στους κανόνες με το σωστή αναλογία πολιτικών και στρατιωτικών μέτρων. Γιατί αυτό αναφέρουν οι συνθήκες και γιατί έτσι θα δημιουργηθεί η ειρήνη. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες του κυρίου Ντανζάν, αλλά θα καταψηφίσουμε την έκθεση αν δεν γίνουν δεκτές τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ριβιέρ για ένα λεπτό. Σε θέματα διπλωματίας, ασφάλειας και άμυνας, ο κύριος Νταζόν και ο κύριος ε, Μακάλιστερ έκαναν καλά δουλειά, τους ακούσαμε προσεκτικά. Βέβαια, δίνουν την εντύπωση ότι πιστεύουν ακόμα λίγο στο έθνος. Ε, παρόλο ότι καταλαβαίνω και συμμερίζομαι κάποιες από τις αναλύσεις τους για το δημογραφικό, για τον Ισλαμισμό κλπ. Ε, δυστυχώς ε, η ε, προσέγγιση τους δεν συνάδει με μια ενωμένη αλληλέγγυα Ευρώπη. Ε, αυτή τη στιγμή η πολιτική μας υποστηρίζει πολύ συχνά προγράμματα αποσυνδεδεμένα μεταξύ τους, που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Ε, η στρατηγική αυτονομία κάθε χώρας έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ζητάει ο κόσμος και με την συνθήκη. Ε, με διάφορες ε, τροπολογίες γίνεται προσπάθεια ε, να προσαρμοστεί η πολιτική της Ευρώπης σε εθνικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε κυρία Φωτίγκα για ένα λεπτό. Thank you. Uh, I focus on... Uh, Ευχαριστώ. Ε, ε, είναι πολλά ε, τα θετικά στην έκθεση, όπως γνωρίζουμε, όπως είναι η ελευθερία ε, της ναυσιπλοείας, προκλήσεις και απειλές ε, σε αυτή την έννοια, από τα στενά του ορμούς μέχρι την Αζωφική θάλασσα. Ωστόσο, βλέπω και κάποιες κόκκινες γραμμές εγώ. Η πλειοψηφία ε, όχι με ομοφωνία, αλλά με η λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία. Α πούμε, στη συζήτηση για το Ιράν είδα ότι είμαστε πολύ διχασμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκτό αυτού, η εισαγωγή της λήψης απόφασης με ενισχυμένη πλειοψηφία μπορεί ε, να είναι εις βάρος της περαιτέρω ενίσχυσης της πολυμερούς συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Γουάλλας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την έκθεση αυτή πρέπει να πω ότι βλέπω μια έντονη επιθυμία της διοίκησης για στρατιωτικοποίηση. Αυτό είναι όμως κατά των συνταγμάτων κάποιων κρατών μελών. Η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία έχει αυξήσει την στρατιωτική συνεργασία και αυτό είναι άμεση απειλή προς την ουδετερότητα της Ιρλανδίας. Με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο που ενθαρρύνει η έκθεση Ε, γίνεται μια κούρσα εξοπλισμών. Σε αντίθεση με την έκθεση αυτή που καλωσορίζει την εφαρμογή του μόνιμου διαρθρωμένου διαλόγου και τη συνθήκη τη Λισαβόνα ε, που έγινε νομικά δεσμευτικό, δεν συμφωνούμε. Ε, αυτό ε, δεν συνάδει με τις εθνικές νομοθεσίες και οι πρόσφατες εξελίξεις στην ΚΕΠΑ απειλούν πάρα πολύ την Ιρλανδική ουδετερότητα. Και ποια ε, είναι λογική πίσω από την ε, έκθεση αυτή και τις τροπολογίες. Και το ελεγκτικό συνέδριο έδειξε ότι δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη με αυτή την τάση στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ο συνάδελφος ε, Ντεμόν για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Κύριε Μπορέλ, ε, ένα από τα μεγαλύτερα ατού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι η ήπια δύναμή μας. Η αξιοπιστία μας ε, στην προστασία, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία, για στην προστασία τους, των μειονοτήτων και της αντιπολίτευσης, δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε. <clears throat> Τι θα πούμε αν η ομάδα εργασία του ΟΕΕ πει ότι μια τρίτη χώρα έχει φυλακίσει εννιά άτομα και θα πρέπει να, αδικά ε, και θα πρέπει να απελευθερωθούν. Θα ήταν ε, εξωφρενικό, θα διαμαρτυρόμασταν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έκανε ισχυρέ δηλώσει ε, εναντίον αυτή τη απειλή. Τι θα γινόταν όμω αν, από αυτές, αν αυτή η χώρα ήταν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν στην Ισπανία. Οπότε θα ήθελα να, να ρωτήσω αν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της δημοκρατικής αξιοπιστίας της εξωτερικής μας πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ζητά τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια που ζητά και από τα υπόλοιπα, μέλη του, υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Και τώρα ακολουθεί η Γκάλ για ένα λεπτό. Το βασικό στόχος ε, της πολιτικής μας είναι και πρέπει να είναι ε, να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία, να προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα, να ανασταλούν οι μεταναστευτικές ροές ε, και να προλάβουμε νέες μεταναστευτικές ροές. Όλα αυτά εντάσσονται στο θέμα που συζητάμε και πρέπει να αποφύγουμε και περιφερειακές συγκρούσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Στην κοινή πολιτική ασφάλειας είναι βεβαίω ευχάριστο το γεγονός ότι θέλουμε να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά μέχρι τότε ε, είτε στα κράτη-μέλη να καταβάλουν προσπάθειες. Παραδείγματο χάρη σε εμά υπάρχει μια, ένα σημαντικό μέτρο για την ανάπτυξη στρατού και ε, πάνω από 2% του ΕΠΑ θα διαθέσουμε για το σκοπό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να εμφανιστούμε και σε άλλες περιοχές, ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Οφείλουμε να συνεργαστούμε με την Αλβανία και τη Βόρεια ε, Μακεδονία. Με την ειδική πλειοψηφία δεν συμφωνώ γιατί αυτό αφαιρεί από τις μικρές χώρες τη δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή τους σε σημαντικά θέματα και να διαφυλάσσουν τα εθνικά οικονομικά του συμφέροντα. Ο κύριος Πίκουλα, παρακαλώ. sigurnosne politike je doneseno konsenzualno. Istaknuta je uloga Evropske unije ne samo u promoviranju aφορά αυτά που είπαν οι συγητές, έχουμε την ε, στάση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, αυτό είναι κάτι επί το οποίο πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Όσον αφορά την ΚΠΑ και την κοινή πολιτική ασφάλειας, ελπίζω αυτή η έκθεση να στηριχθεί στο μέλλον, όπως επίσης και οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τις πρώτες εβδομάδες αυτού του έτους είδαμε ότι στην περιοχή υπήρξε συμβολή στη σταθερότητα. Γι' αυτό και θελήσαμε να προάγουμε τις βασικές αξίες της ε, Ειρηνή και της συνεργασία. Ε, στρατηγική λοιπόν αυτονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει τις δυνατότητες της ε, άμυνας. Εγώ πιστεύω ότι τα Βαλκάνια θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική ασφάλεια. Μια σταθερή πολιτική είναι μια εγγύηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά είναι τα μηνύματα που πρέπει να στείλουμε ε, στους εταίρους μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ισχυρή Ευρώπη ε, σε ένα κόσμο πολυμερών σχέσεων. Ε. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η κυρία Ναταλή Λουαζό από την ομάδα ΡΕΝΙΟ η κυρία Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μια γεωπολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει δίκιο αυτό, το δείχνει η κατάσταση του κόσμου. Στην άμεση γειτονία μα βλέπουμε ε, που τραβάνε σε μακρο και ε, σε πλάτο και σε χρόνο. Οι κρίσει πολλαπλασιάζονται, διαιωνίζονται ε, και θα πρέπει να ξεφύγουμε από τα χρόνια της αθωότητας όπου το ευρωπαϊκό εγχείρημα ήταν ε, εγχείρημα ειρήνης και δεν ήταν η άμυνα αυτό που το ενδιέφερε από την ξενιασιά του. Ε, τώρα χαιρετίζω την έκθεση που ε, θυμίζει τη σημασία ε, της συμμαχίας μας και της πολυμερούς αποτελεσματικής συνεργασίας, αλλά καλή στη δημιουργία μιας βαρύς ευρωπαϊκής άμυνας για να μπορέσουμε να ανταποκρινόμαστε από τη μια στις δεσμεύσεις απέναντι στους συμμάχους, αλλά να έχουμε και αυτόνομη δραστηριότητα κάθε φορά που το απαιτούν τα συμφέροντά μας. Είναι διακαής ανάγκη πλέον αυτό. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κατηγορούμε τους Αμερικανούς συμμάχους μας ότι το παρακάνουν ή ότι δεν κάνουν αρκετά σε κρίσεις ή περιφέρειες που άμεσα μας αφορούν. Θα πρέπει να αναλάβουμε όλο το μερίδιο που μας αναλογεί και στην πρόληψη των κρίσεων αλλά και στην επίλυσή τους. Χρησιμοποιούμε όλα ε, τα εργαλεία Προ το σκοπό αυτό. Ας είμαστε διαμεσολαβητέ, διευκολυντέ, αλλά και πρωταγωνιστές ε, στην ειρήνευση όταν διακυβεύονται τα δικά μας συμφέροντα. Θα πρέπει να ε, δεχθούμε ότι θα βαρύνουμε με όλο το πολιτικό βάρος που μας δίνει η οικονομική μας ισχύ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε πλέον σε άλλες δυνάμεις ε, τη φροντίδα να διαμορφώνουν το γεωπολιτικό μας περιβάλλον χωρίς να ακούγεται η δική μας φωνή. Η Ευρώπη ε, έχει συνηθίσει να μιλάει και να κουβεντιάζει και τώρα έχει έρθει η ώρα να δράσει. Για ένα λεπτό ο κύριος Ντεμάν από την ομάδα ε, Ταυτότητα και Δημοκρατία. Πολλά ακριβά λόγια ακούμε και ωραίες αρχές, αλλά κυρίως ε, πολλές αερολογίες. Η χειρότερη άμυνα για την ασφάλεια, μάλλον για την